Συνεχίζεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά τη πεσινής συνεδρίαση σα έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, ε, η έγκριση των πρακτικών ε, είναι δεδομένη. Στην ημερήσια διάταξη τώρα έχουμε την δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής